Ε, ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Ε, θα ήθελα να αρχίσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Παρακαλώ να σταματήσουν οι παράλληλες συζητήσεις. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Έχετε βάλει στις χισμές τις κάρτες σας. Και μπορούμε να κάνουμε μια δεικτική δοκιμαστική ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι για τρεις ώρες ψηφοφορίας. Αρχίζει η ψηφοφορία, δηλαδή η δοκιμαστική ψηφοφορία. Ευχαριστώ πέρας. Καταπληκτικό. Η πλειοψηφία είναι έτοιμη για να ψηφίσουμε τρεις ώρες, θα, στη μία θα ολοκληρώσουμε. Διαδικαστικό ταμπουράνο. Ε, Γεια σας Πρόεδρε, γεια σας συνάδελφοι. Λαμβάνοντας υπόψη την περιπλοκότητα της ψηφοφορία για την Ενεργειακή Ένωση και τα πολλά σημεία σημαντική σημασία. θα ζητούσα από, τον Πρόεδρο στο τέλος της ψηφοφορία, μάλλον μετά την τελική ψηφοφορία επί της εκθέσεως, ε, ε, να σταματήσουμε για 5-10 λεπτά έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, αποφασίσουμε, να δούμε ποιο είναι το κείμενο τελικά έτσι όπως θα έχει ψηφιστεί. Να σταματήσουμε, να κάνουμε μια διακοπή για 10 λεπτάκια. Ναι, εντάξει, αλλά θα, ε, δεν θα έχουμε χρόνο. Δύο-τρία λεπτά, όχι παραπάνω. Να είστε έτοιμοι για αυτή τη ε, διακοπή, αλλά όχι 10 λεπτά. Κανονικά είναι 2-3 ε, λεπτά πριν τελική ψηφοφορία. Λοιπόν, Επιλέξιμη υποψήφοι για το διορισμό στη θέση του των εκπροσώπων συγγνώμη, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Acer. Η Ρωμάνα Γιόρνταν είναι η υποψήφια μας. Ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. συγγνώμη, δύο υπεράριθμοι ΕΛΚ. Περισσεύουν δύο από το ΕΛΚ. Ωραία τώρα, πολύ ωραία. Πέρας ψηφοφορία, ευχαριστώ. Ούβε τώρα, αναπληρωτής, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Ωραία. Πέρασε η πρόταση. Τώρα θα ψηφίσουμε για τον κατάλογο των υποψηφίων, για όλους μαζί. Χρειαζόμαστε την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ήτρε. Άρχεται ψηφοφορία για τον κατάλογο, για ολόκληρο τον κατάλογο των υποψηφίων. Πέρας. ΕΛΚ. Περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Τώρα εντάξει. Πέρας. Πολύ ωραία. 55 ψήφοι υπέρ ε, και 6 αποχές. Θετική έκβαση της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια στους ε, υποψηφίους μας θα διοριστούν από την διάσκεψη των Προέδρων. έκθεση για το, 10, το στόχο του 10% για την διασύνδεση των ε, δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος. Συνάλφος Έριξον. Συμβαστική ένα υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, συγγνώμη, μείον ένα με αρνητικό πρόσημο. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική ένα τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά τμήματα είναι. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Το δεύτερο τμήμα της 22. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απερίφθη. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έλεγχος. Για την 57 έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 76. 76. Ηλεκτρονικά. Πέρας. 76. Πέρας. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 7α υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 77 έλεγχος. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πάλι έλεγχος. Για την 78. Περισσεύει ένα σέλκ. Τώρα εντάξει. Πέρας. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, για την 90 θέλετε έλεγχο. Όχι. Για τη συμβαστική λοιπόν, ε, ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται κατά πασαφθενότητα, αλλά έλεγχος παρακαλώ, 106. 106. Πάλι περισσεύει κάποιος από το ΕΛΚ. Ένας. Ευχαριστώ. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, συμβαστική 17 υπέρ κατά συμβαστική εγώ έκανα λάθος λέω πρώτος συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική μείον 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έτσι δεν είναι έλεγχος 167 167 πέρας εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 20α υπέρ 168 καλά οκ okay. 168 ε, ε. εγώ τι είπα εγκρίθηκε απορρίφθηκε ζητώ συγγνώμη επανάληψη 168 ψηφίστε και πάλι παρακαλώ 168 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, δίκιο είχα. Καλά το είπα ότι απορρίπτεται. Πρώτη φορά το πέτυχα. 20α ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική 22 187. 187 έλεγχος πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 ε, υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Συμβαστική 22. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τώρα, τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την τροπολογία 1. Για την τροπολογία 1 κάνουμε έλεγχο. Σημαστική. Α, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική, ονομαστική. Άρχεται. Πέρας. Α, πάλι περισσεύει κάποιος ΕΛΚ. Πέρας. Ευχαριστούμε, συγχαρητήρια. Ε, Σνάλφε Έριξον. Πάμε τώρα στην... επόμενη. Ε, σχέδιο έκθεσης για μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Εισηγητής ο κύριος Γκρομπάρτζικ. Point of order, Point Επί τη διαδικασίας, ο κύριος Γκρομπάρτσικ. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία που είχαμε ειδικά τους κοιόδης εισηγητές όλων των ομάδων. Κάποια πράγματα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά για να σεβαστούμε τις ε, κόκκινες ε, γραμμές όταν μιλάμε για στόχους. Οι συμβαστικές 67β 26B 26B 263 και 265 είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς δηλαδή το να απορριφθούν γιατί για το ECR αυτά είναι κόκκινη γραμμή και θα μας αναγκάσουν να καταψηφίσουμε όλη την έκθεση και σας παρακαλώ να σεβαστείτε τη θέση μας. Σας ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Κύριε Τούρμας, τώρα δεν είναι η ώρα για να μπούμε στην ουσία. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα είναι σημαντική για την κλιματική αλλαγή, για την παραγωγικότητα της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας για ανεξαρτησία από ανθρώπους όπως ο κύριος Πούτιν οπότε νομίζω πως λογικό είναι να ζητάμε στιβαρούς στόχους για την αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ κύριο Σταμπουράνο. Εγώ δεν πιστεύω πως ε, τώρα εδώ πέρα είναι η στιγμή για να πούμε ε, να ψηφίσουμε ή όχι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα κανονικά με την ε, ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση κύριε Σιγητά να σας συγχαρώ γιατί θα γίνεται μάλλον μέλος της πολωνικής ε, κυβέρνησης μαζί με τον άλλον συνάδελφο τον κύριο Γεσκεβίτς και, και από ό,τι φαίνεται και ο κύριος Σιμάνσκι ε, τον οποίον επίσης ε, θα θυμάστε ότι ήταν μέλος της Επιτροπής μας. Μιλάμε για κυβέρνηση Ήτρε στην Πολωνία. Συγχαρητήρια συνάδελφοι. Τροπολογία 2.49 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας. Απορρίπτεται. 2.50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.52 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2.56 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή ένβη 48 υπέρ κατά αποχές 10.16 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.63 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 2.65 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 2.65 λοιπόν Πέρας. Απορρίπτεται. 2.66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 2.66. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται όμως 264 264 πέρας δεκτή ωραία δύο μαζί κατόπιν 251 και 267 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές ε, δεκτές συμβαστική τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή 4.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εντάξει 4.50 πέρας απορρίπτεται τα 21 υπέρ. Κατά. Πρέπει να την επαληθεύσουμε. τα 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 2.85 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.97 υπέρ κατά αποχές δεκτή μάλλον α την επαληθεύσουμε εντάξει 2.97 2.97 πέρας δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7.30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6.37 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή άφετ 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή άφετ 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή άφετ 15 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.43 υπέρ. Κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 3.43 πέρασε απορρίπτεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 β υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, ωραία 13β άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται συμβαστική 30 καλά κάναμε λοιπόν και τα παληθεύσαμε 13α υπέρ κατά αποχές δεκτή 4-15 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 4-15 πέρας απορρίπτεται 4-16 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 447 υπέρ κατά αποχές δεκτή ωραία να τα παληθεύσουμε 447 447 πέρασε Δεκτή. 4.32 υπέρ κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε και αυτήν. 4.32 Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προσθήκη ένα υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε την προσθήκη 1 παρακαλώ πέρας δεκτή προσθήκη 2 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε και πάλι προσθήκη 2 πέρας δεκτή 486 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε και πάλι 486 να την επαληθεύσουμε πέρας δεκτή 17α υπέρ κατά αποχές δεκτή ίντα 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται ε, να 13 ναι, υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε πέρας δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε και αυτήν την 16 αρχη τη ψηφοφορία πέρας δεκτή νομίζω είναι τα 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή να την επαληθεύσουμε όμως άφετ 10 Αυτήν ψηφίζουμε. Και πέρας. Δεκτή. 4,97 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5,04 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5,02 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται εντάξει εντάξει να την επαληθεύσουμε 5-0-2 5-0-2 πέρας δεκτή δεκτή ναι, έχετε δίκιο σας ευχαριστώ 5-0-6 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 5-0-6 Πέρας. Δεκτή. 5-0-3 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορριπτεται 5 5-0-0 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4-99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. δεκτη Δεκτή. 5-0-1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ψηφίσατε καθόλου. 501 και πάλι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 507 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 507. Να την επαληθεύσουμε. Πέρες. Δεκτή. 793 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 5 1-1 5-11 δηλαδή υπέρ κατά αποχές δεκτή 10-50 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 1-0-5-0 πέρασε Δεκτή. 5-1-3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5-1-5 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5-17 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. 5-17 επαληθεύουμε την 517. Πέρας. Απορρίπτεται, μάλιστα. 519 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε, παρακαλώ. 519. να την επαληθεύσουμε, ναι, ναι. Λοιπόν, πέρας δεκτή συμβιβαστική 18 α 5-16 5-16 5-16 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε και πάλι 5-16 πέρας δεκτή Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 5.26 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 5.21 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 5.23 υπέρ. Κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 5.23 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 5-29 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 569 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 573 υπέρ κατά αποχές δεκτή 574 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 574 πέρας δεκτή 5.75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε και πάλι. 5.75. Πέρας. Απορρίπτεται. 5.65 πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6-20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 21β υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 21β πέρας απορρίπτεται 21α υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6.47 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 6.47 πέρας δεκτή 3.01 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 301 Δεκτεί. δεκτή άρα 6.33 μέρος πρώτο εκεί πάμε λοιπόν στο πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 6.33 μέρος πρώτο πέρας υπέρ 6.29 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 629. Πέρας. Δεκτή. Συνάδελφοι, σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ γιατί αλλιώς δεν βλέπω. Ε, 8.52 υπέρ. Κατά. Αποχές να την επαληθεύσουμε. 8.52 την επαληθεύσουμε πέρας δεκτή 6.38 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε και αυτή δεν σηκώνται τα χέρια λοιπόν να την επαληθεύσουμε 6.38 Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 26 υπέρ. 23, 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συγγνώμη, συγγνώμη, διάλειμμα. It's um, nothing with alcohol. It's... Um, <laughs> ε, δεν πίνω ινόπνευμα πρωί-πρωί. You can check if anybody wants. Άμα θέλετε, ελάτε να δείτε. Όχι, όχι ηλεκτρονικά όμως. Λοιπόν, 6, 6, 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαλτεύσουμε. 6, 6, 7. Πέρας. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έξι έξι υπερ Κατά. Αποχές. Έξι εφτά μηδέν υπερ Κατά. Αποχές. Να την απολυθέψουμε. 6.70 λοιπόν 6.70 πέρας απορρίπτεται η 6.70 υπέρ 6.72 ε, με συγχωρείτε υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 6.72 την επαληθεύουμε πέρας Δεκτή. 6,77 υπέρ. Κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 6,77. 6,77. Πέρας. Δεκτή. 6,75 υπέρ. Κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 6.75 πέρας δεκτή 6.80 υπέρ 6.80 υπέρ κατά αποχές δύσκολο να την επαληθεύσουμε λοιπόν. Πέρας. Δεκτή. 6-8-8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 6-84 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 6-85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1160 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1161 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 1161 πέρασε 6, 8, 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 8-0-6 υπέρ υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. ΕΜΕ έχει γίνει δεκτή. Α, με συγχωρείτε. 8-0-6, 8-0-6 είχε γεννιδεκτεί. Άρα περνάμε όχι στη συμβαστική 24, αλλά στην τροπολογία 6 23, 6 23, 3 6-2-3 μετα την 8-0-6. 623 υπέρ κατά αποχές δεκτή τώρα πάμε στη συμβαστική 24 βιάστηκα λίγο Συμβιβασμός 24 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 693 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7, 27, 7, 27, 24. Τμήμα 2. Όλα αυτά είναι ταυτόσημα. Τέσσερις τροπολογίες από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 891 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 726 υπέρ κατά αποχές να ε, ελέγξουμε 726 ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 726 πέρας δεκτή 7.25 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5.50 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 562 υπέρ 562 562 ε, το 550 εγκρίθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι η είναι καταπίπτει και επομένως ψηφίζουμε την 562 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 563 υπέρ. Κατά καλύτερα να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση 563. 563. Πέρας. Απερίφθη. 553 υπέρ κατά αποχέσε απερίφθη 555 υπέρ κατά αποχέσε εγκρίνεται Πηγαίνουμε στην τροπολογία 732 υπέρ κατά καλύτερα να ελέγξουμε. Επαλήθευση λοιπόν επί της 732. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απερίφθη. 733 υπέρ. Κατά. Αποχές πάλι να ελέγξουμε. Επαλήθευση λοιπόν από τις 7.33. 7.33 ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρας, απερίφθη. Συμβιβασμός 26B, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση είναι πολύ σημαντικό. 26Β, Πέρας. Απερίφθη. 26α ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 είναι πάντα συμβιβασμοί συμβιβασμός 27 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 790 υπέρ κατά αποχές νομίζω πως εγκρίθηκε αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε 790 790 ηλεκτρονική επαλήθευση πέρας ε, ναι είναι αποδεκτή 794 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 807 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία 811 ε, υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 8.11 επί 8 8.11 πέρας απερίφθη 808 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 810 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβασμός 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV29 υπέρ κατά NV28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 855 υπέρ κατά αποχές καλύτερα να επαληθεύσουμε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 855 πέρας της ψηφοφορίας. Αποδεκτή. Τροπολογία 812 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 859 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, συμβιβασμός 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 32 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 881 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 881. 881 πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη συμβιβασμός 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 922 υπέρ κατά καλύτερα να κάνουμε την επαλήθευση επί της τροπολογίας 922 Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη υπέρ. Κατά. Καλύτερα να ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την προσθήκη πέρας της ψηφοφορίας Αποδεκτή. Τροπολογία 941 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 942 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 971 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση 971. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ένβη 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ένβη 40 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εν... 41 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να ελέγξουμε 42 ηλεκτρονική επαλήθευση NV42 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 55 NV υπέρ κατά αποχές καλύτερα να ελέγξουμε για μια ακόμα φορά NV55 άρχεται η ψηφοφορία πέρας αποδεκτή Συμβιβασμός 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. nv 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά ε, να ελέγξουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την NV25. Πέρας. Απερίφθη. Συμβεβασμός 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός... Τι λέτε... Ναι, είμαι συμβιβασμό 35. Εγώ νομίζω ότι ήταν σαφέ το αποτέλεσμα, αλλά να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Πέρας. αποδεκτή τροπολογία ε, συμβιβασμός 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προσθήκη 1 υπέρ κατά αποχές ε, καλύτερα να επαληθεύσουμε πέρας απερίφθη προσθήκη 2 υπέρ κατά αποχές, νομίζω και αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Προσθήκη 2 λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Αυτή τη φορά αυτή η προσθήκη γίνεται δεκτή. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 897, 897 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση 897. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 703 υπέρ. Κατά. Ε, και πάλι έλεγχος 703. Ε, Πέρας ψηφοφορίας για την 703 εγκρίνεται, εγκρίνεται αυτή τη φορά. 11-19 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11-20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11-21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 977 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Τώρα 982. Ναι, 982. Γιατί εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα και πρέπει να πάμε στο 982. Σωστά. Το πρώτο τμήμα της 982 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. 982 πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά έλεγχος έλεγχος για να είμαστε σίγουροι πέρας εγκρίνεται τώρα Το τρίτο τμήμα. Α, εννοείται επειδή ήταν τρίτο τμήμα πριν. Άρα καταπίπτει το τρίτο τμήμα ουσιαστικά. 983. 983 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. 983. Συνάδελφοι, είναι περίπλοκο. Πρέπει να προσέξουμε τι κάνουμε. 983. Πέρας. Απορρίπτεται. 975 υπέρ κατά Έλεγχο, παρακαλώ 975 πέρας εγκρίνεται 980 πρώτο τμήμα 980 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα κατά αποχές Εφτά. 3 Ένα. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, προσθήκη υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την προσθήκη ονομαστική ψηφοφορία φυσικά ηλεκτρονική Έλεγχο έλεγχος παρακαλώ πέρας ωραία εγκρίνεται 9-9-6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1002 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 992 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. 992. Πέρας ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 9-5 ναι, ναι, υπέρ. Κατά. 9.95 έλεγχος. Πρέπει να γίνει έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 9.93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 998 υπέρ κατά έλεγχος έλεγχος 998 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1003. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1001 υπέρ κατά απο, αποχές έλεγχος πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 1000 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Έλεγχος για την ε, τροπολογία 1000. Πέρας. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Πρέπει να γίνει έλεγχος για την 997. 9, 9, 7. Πέρας. Απορρίπτεται. 1004. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1015 υπέρ κατά πρέπει να γίνει έλεγχος 1015 Πέρας. Εκρίνεται. Τρεις θέσεις μαζί πρέπει να ψηφίσουμε. Την 1017, τη 1018 και την ναι, 1019 καθώς και την 1020. Αυτές τις τέσσερις τροπολογίες είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. 1026 υπέρ. Ε, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, ένα λεπτάκι. Ναι, εγκρίθηκαν. 1035. Συναδελφοί, ε, δεν έχω κανένα ανέκδοτο να σας πω για να χαλαρώσουμε λίγο, αλλά ας πάμε στη 1035. 1035, υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 1035 όπως λέγαμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 1037 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να κάνουμε έλεγχο. 1037. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 1037. Πέρας. Εγκρίθηκε πολύ ωραία. Τραν 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τραν 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1038 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 14 την επόμενη σελίδα. Τραν 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τραν 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχε... αποχές έλεγχος παρακαλώ Συ... συνάδελφοι παρακαλώ μην κατεβάζετε τα χέρια τόσο γρήγορα γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τραν 13 έλεγχος Άρχεται, πέρας, περίφθη. MV37, 36 ε, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. MV37 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1048 υπέρ κατά Αποχές... Ε, α, έλεγχος, καλά, 1048, έλεγχος. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 317 17, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 315 Κατά αποχές εγκρίνεται, 1051 και 1052 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες. Ε, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ε, συμβασμό 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε, προσθήκη υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. την προσθήκη για τη συμβαστική 40 ψηφίζουμε πέρας. Πέρα, απορρίπτεται. Συμβαστική 241 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 1, ε, ε, προσθήκη 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη 2 για τη συμβαστική 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη 3 υπέρ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 11-24 υπέρ. Αν θέλετε ε, να ελέγξουμε την προσθήκη 3, κανένα πρόβλημα. Καλά. Προσθήκη 3. Προσθήκη 3. Πέρας εγκρίθηκε 11.24. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8.65 υπέρ. Κατά. Έραγχος. 8.65. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. MV39 υπέρ. Κατά. Πρέπει να το ελέγξουμε. MV39. Εγκρίθηκε. Πέρασε. Συνάδελφοι, ξέρω ότι έχετε κουραστεί, αλλά πρέπει να σκόνετε τα χέρια, αλλιώς δεν μπορώ να μετρήσω. Εγκρίνεται. 1100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11.02 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11.06 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11.01 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11.09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1.1.2.3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1.1.2.9 υπέρ Κατά. Έλεγχος για την 1129. Πέρασε. Εγκρίνεται. 11, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11.34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11.44 υπέρ έλεγχος καλά 11.34 έλεγχος Πέρας. Εγκρίνεται. 11.44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να γίνει έλεγχος. Παρακαλώ. 11.44. Πέρας. Δεκτό. 11.48 υπέρ. Κατά. Είναι. 11.48. Πέρας ψηφοφορίας. 11.49 υπέρ. Κατά. Και αυτός εδώ έλεγχος. 11.49. Πέρας. Εγκρίνεται. 11.56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11.62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 2. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Έλεγχος για τη 2.14. 2.14. Close the vote. Is rejected. Απορρίπτεται. Μαζί δύο τροπολογίες ταυτόσουμε στις 45 και οι 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος. 45-47. 45-47. Μαζί. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 67. Το δεύτερο τμήμα. Δεύτερο. Συμβαστική. 67. Ε, ε, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Let us check it. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 67 τμήμα 2. I close the vote. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, δεκτή. Τροπολογία 69. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 71. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 50 ή μάλλον όχι, τροπολογία 82 πρώτα. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 86 υπέρ κατά. να ελέγξουμε τροπολογία 86 ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, τροπολογία 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 109 τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 Υπερκατά κατά, αποχές, εγκρίνεται. αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Επαλήθευση λοιπόν επί της τροπολογίας 130. Τροπολογία 130. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 54. Ε, Υπερκατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 100, τροπολογία 138, 138 υπέρ, κατά ε, ηλεκτρονική επαλήθευση 138 πέρας εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δύο τροπολογίες μαζί, η 140 και η 141 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση επί δύο ταυτοσύμων τροπολογιών 140-141 επαλήθευση πέρας εγκρίνονται τροπολογία 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 142 142 πέρας απερίφθη 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά. Τι να σας πω, δεν είναι σαφές. 144 ηλεκτρονική επαλήθευση. 144. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 147 και 148 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω αλλά καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση 176 πέρασε Απερίφθη. 175 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε, αλλά νομίζω ότι απερίφθη. 175 ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασε. Α, και όμως γίνεται δεκτή. 177. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έξι τροπολογίες μαζί, 155, 156, 157, 158, 159, 160 είναι ταυτόσιμες και τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στην τροπολογία 172 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για την 173. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 57 υπέρ κατά. «57 ηλεκτρονική επαλήθευση, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν, πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 136 υπέρ. Κατά. Ε, να ελέγξουμε καλύτερα. 136. Πέραση της ψηφοφορίας. Απερίφθη. Συμβιβασμός 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 184 υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση επί της 184. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. 185 υπέρ. Κατά. Απερίφθη, αλλά καλύτερα να το τσεκάρουμε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση 185. Πέρας. Απερίφθη. 186 υπέρ. Κατά. Η ίδια πλειοψηφία απερίφθη. 187 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 188 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 189 υπέρ κατά ε, Τώρα είναι λίγο διαφορετικό το αποτέλεσμα, ίσως έγινε δεκτή η τροπολογία αυτή, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της 189. Πέρασε. Δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα στην τροπολογία 243. 243. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβιβασμός 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 200 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά ε, να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 2.16. Πέρας. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι πάμε στο συμβιβασμό 60. Η υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 242 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 246 υπέρ, κατά. Να κάνουμε την επαλήθευση επί της 246, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. απερίφθη απερίφθη. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Όχι, όχι, το συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 απορρίπτεται, τροπολογία 2 εγκρίνεται. Τροπολογία 3 και 4 είναι ταυτόσιμες, τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ 12 10 και 12 μαζί λέει ο πρόεδρος τώρα είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 υπέρ κατά να ελέγξουμε τροπολογία 13 ηλεκτρονική επαλήθευση Πέρας της ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Ε, δύο τροπολογίες μαζί, τροπολογία 14 και τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και οι δύο Επομένω είναι δεκτές τροπολογία 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, καταλαβαίνω ότι τώρα θέλετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, δύο-τρία λεπτάκια αγαπητοί συνάδελφοι.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 Uh, uh, and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, τώρα είμαστε απολύτω έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι νομίζω για την τελική ψηφοφορία. Ε, θα γίνει με ονομαστική κλίση. Σας παρακαλώ να καθίσετε στις θέσεις σας και να ψηφίσετε. Αρχίζουμε λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία για την τελική ε, ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 47 ψήφοι υπέρ, επομένως ε, να ε, συγχαρούμε τον Στάνφερ Κουμπάτσικ και όλους τους σκιώδεις. Ήταν πολλές οι τροπολογίες, πολλή δουλειά, πολύ σκληρή δουλειά των ε, σκιωδών αλλά και του εισηγητού φυσικά και επομένως περνάμε ε, στην τελική ψηφοφορία για το επόμενο θέμα Corporate Tax Policies Μασιμιλιάνο Σολίνη είναι ο εισηγητής μας και να ξεκινήσουμε λοιπόν Συμβιβαστική τροπολογία 1 με τις προφορικές τροπολογίες της ΑΛΤΕ Κυρία Κάλλας ε, έχει ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας Έχετε προφορική τροπολογία. Μάλιστα, ναι. Εξ ονόματος της ΑΛΔΕ θα ήθελα να προτείνω μια προφορική τροπολογία 1 στο 1α να αντικατασταθεί η προσεκτική αξιολόγηση με αξιολόγηση αντικτύπου γιατί η προσεκτική αξιολόγηση δεν υπάρχει στο ευρωπαϊκό δίκαιο οπότε ζητάει να ξαναξεκινήσει η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση και ζητάει την ε, πλήρη εφαρμογή της ε, με βάση μια συνολική αξιολόγηση αντικτύπου κτλ. Any, any objections? Υπάρχει αντίρρηση. Πρέπει να σηκωθείτε αν έχετε αντίρρηση. Όχι. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε μια συμβαστική τροπολογία μαζί με την προφορική τροπολογία της κυρίας ε, Κάλλας. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 13 χωριστή ψηφοφορία μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά δεν σηκώνεται το χέρι πώς να καταλάβω να την, να την επαληθεύσουμε. Τροπολογία 15. Να έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 31 υπέρ δεύτερο μέρος δεύτερο μέρος είναι για το πρώτο καταπίπτη μέρος 31 δεύτερο μέρος υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε. Τροπολογία 31, δεύτερο μέρος. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ συμβιβαστική. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε 48 πέρας δεκτή Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογική 62 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. 62 ε, ηλεκτρονική επαλήθευση πέρασε απορρίπτεται 63 σε τρία μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε μέρος πρώτο της 63 πέρασε δεκτή δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος τρίτο υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε 73 73 Πέρας. Δεκτή. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Να, να την ξαναδούμε. 75. Μάλλον δεκτή. Για να δούμε. Πέρας. Ναι, παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. Δεκτή. 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 σε δύο μέρη 81 81 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 81 μέρος πρώτο Καλησπέρα. Απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται επίση. Τροπολογία 83 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. 83. 83. Επαληθεύουμε τον 83. Πέρασε. Δεκτή. 85 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 86 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 87 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχίτη ψηφοφορία. Πέρας. 49 υπέρ Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη. Μια μισή ώρα τα καταφέραμε και ήσασταν προετοιμασμένοι και για τρεις ώρες. Τι να κάνετε, πήγαινε για... να φάτε. Ναι. Commissioner stays Συνάδελφοι, στην ημερήσια διάταξη έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Την ε, διαπραγμάτευση για την TTIP, την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου. Οπότε καθίστε μαζί μας γιατί μέχρι τη μία η ώρα είμαστε ελεύθεροι. Dear colleagues, uh, if you cannot stay with us, please. Αδελφοί, παρακαλώ όσοι δεν θέλουν να αποχωρήσουν ήσυχα. Quick as possible and give us possibility to discuss the next point. Παρακαλώ λοιπόν να μας δώσετε να αποχωρήσετε ήσυχα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Κύριε Τούρμες, ε, κύριε Τούρμες, σας βλέπω ακριβώς μπροστά μου. Θέλουμε να ξεκινήσουμε λίγο τη συνεδρίαση. Συνάδελφοι. Συνάδελφοι εκεί, οι σοσιαλδημοκράτες. Άνταμ, πες, πες τους συναδέλφους κάτι. Κυρία Τόιερ, καθίστε σας παρακαλώ. Λοιπόν, συνάδελφοι, διαπραγματεύσεις TTIP, Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων. Καλωσορίζω τον κύριο Πέτρο μέλη επικεφαλής έρευνας αγοράς ε, στην DigiTrade. Ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή μας και αναμένουμε την ενημέρωσή σας για τον 11ο γύρο συνομιλιών που έλαβαν χώρα στο Μαϊάμι 13 με 17 Ιουλίου. Οι διαπραγματεύσεις να σας υπενθυμίσω ξεκίνησαν επισήμως τον Ιούλιο του 2013. Είμαστε λοιπόν μετά από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων 11 γύρους ο τελευταίος στο Μαϊάμι να σας υπενθυμίσω επίσης πως πέρα από τις επίσημες διαπραγματεύσεις ε, έχουν γίνει και τα εξής ε, μετά την τελευταία ενημέρωση από την Κομισιόν στην Επιτροπή Ήτρα. Πρώτα απ' όλα, αγαπητοί φίλοι, σας παρακαλώ. Ησυχία. Η Επίτροπος ε, Σεσίλια Μάλμστρομ συναντήθηκε με τον κύριο Μάικλ Φρόμαν απεσταλμένο για το εμπόριο των ΗΠΑ για να γίνει μια ανασκόπηση των διαπραγματεύσεων TTIP και στις 5 Οκτωβρίου 2015 η ΕΠΑ μαζί με 11 άλλες χώρες ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία του ειρηνικού η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί. Μας είπαν πως η εμπορική συμφωνία ΕΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει παγώσει από την πλευρά των ΕΠΑ λόγω των επιταχυμένων διαπραγματεύσεων με τον ειρηνικό. Και η Επιτροπή θα ήθελε να ακούσει αν τα συμπεράσματα ε, του TPP έχουν ήδη ε, κάποιο αποτέλεσμα στις συζητήσεις ε, TTIP με τροποθετικό ή αρνητικό. Πώς το βλέπετε αυτό το πρόβλημα. Γιατί για εμάς είναι ανοιχτό. Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία του Ειρηνικού πριν από λίγες εβδομάδες και ίσως έχουμε το επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Καλημέρα και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας καλέσατε να σας ενημερώσουμε για τον τελευταίο γύρο της ε, TTIP. Πριν από δύο εβδομάδες έλαβε χώρα, 9-12 Οκτωβρίου έγιναν συναντήσεις στην Ουάσιγκτον, αλλά πράγματι περισσότερο ήταν στο Μαϊάμι. Ο ενδέκατος αυτός ε, γύρος ε, ήταν ένας καλός γύρος, δουλέψαμε σκληρά και είχαμε κάποια πρόοδο και ένταση των συνομιλιών σε πολλούς τομείς. Θα έλεγα πως τα σκαϊτανισδήματα δήματα πρόσβασης αγοράς είχαμε μία ανταλλαγή αναθεωρημένων προσφορών δασμών και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα συγκρίσιμο επίπεδο όσον αφορά την κάλυψη των δασμολογικών γραμμών, ένα 97% που καλύπτονται από τις προσφορές και είναι θα έλεγα ισορροπημένες με τις αρχικές προσφορές είχαμε μια ανισορροπία με την ευρύτερη κάλυψη που προτείνεται από την πλευρά των ΙΠΑ και ακριβώς τώρα θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η ανισορροπία με τις αναθεωρημένες δασμολογικές ε, προσφορές. Επίσης ανταλλάξαμε προτάσεις με τη ΣΥΠΑ για συγκεκριμένους κανόνες προέλευσης προϊόντων, κάτι το οποίο επίσης είναι σημαντικό, καθώς θα καθορίσει πώς θα ωφεληθούμε από τις ε, προτιμήσεις που θα περιέχονται στην συμφωνία. Μετά, ο δεύτερος πυλώνας μετά τους δασμούς είναι οι υπηρεσίες, και εκεί πέρα ήδη είχαμε αναθεωρημένες ε, προσφορές τον Ιούλιο και εκμεταλλευτήκαμε τον γύρο αυτό για να εμβαθύνουμε τις συζητήσεις και να δημιουργηθεί κάποια πρόοδος ε, όσον αφορά την ενοποίηση των κειμένων. Και ο τρίτος ε, πυλώνας αφορά βεβαίως τις δημόσιες προμήθειες, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ένωση και εκεί πέρα ακριβώς ε, ο γύρος είχε στόχο την προετοιμασία των αρχικών προσφορών και των δημοσίων προμηθειών που είχε προγραμμαστεί για τον Φεβρουάριο. Ο πρόεδρος Μπούζεκ αναφέρθηκε στην ε, συνάντηση των επιτρόπων των, της κυρίας Μάνστρομ με τον κύριο Φρόμαν και εκεί πέρα ακριβώς συμφωνήσαμε στην ανταλλαγή προσφορών για τις δημοσίες προμήθειες μέχρι τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Για να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή. Και βεβαίως και πάλι η πρόσβαση στις αγορές ήταν το βασικό σημείο και βεβαίως είχαμε τα τρία στοιχεία, τους δασμούς, υπηρεσίες και δημόσιες προμήθειες. Βεβαίως είχαμε και άλλες συζητήσεις όσον αφορά την ε, ρυθμιστική διάσταση και συζητήσεις για τους διάφορους κλάδους ε, στους οποίους ε, συζητάμε ακριβώς αυτά τα ρυθμιστικά προγράμματα και τα παραρτήματα. Προφανώς συζήτηση αυτή δεν επηρεάζει ούτε το επίπεδο προστασίας που υπάρχει στους αντίστοιχους κανονισμούς, ούτε ρυθμίζουμε ε, την πολιτική που ακολουθεί του μετά. Στον τομέα των κανόνων, μια σημαντική εξέλιξη ήταν το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε την πρότασή της που είχε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του γύρου και υπήρχαν κάποιες αρχικές συζητήσεις μετά την κατάρτιση της πρότασης της Κομισιόν. Οπότε συζητήσαμε όλα αυτά τα ζητήματα κατά τη διάρκεια του γύρου. Ένα ζήτημα το οποίο δεν συζητήθηκε αφορούσε την προστασία των επενδυτών. Όπως ξέρετε η Κομισιόν έχει κάνει κάποιες σχετικές προτάσεις, αλλά κατά τη διάρκεια του γύρου οι προτάσεις αυτές ήταν σε μια διαδικασία συζήτησης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη, οπότε το ζήτημα αυτό δεν συζητήθηκε. Αυτή είναι η γενική εικόνα, εάν θέλετε, Τώρα, κάποια ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα την Επιτροπή σας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενέργεια και πρώτες ύλες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζετε ότι συζητάμε την συμπερίληψη ενός κεφαλαίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ και θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε τέτοιο κεφάλαιο σε μια εμπορική συμφωνία και κατά τη διάρκεια αυτού του γύρου συζητήσαμε δύο πτυχές την θεσμική διάσταση και βεβαίως ε, τις ε, πληροφορίες και το ζήτημα της συνεργασίας για ζητήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι κάτι στο οποίο έχουμε ήδη συμφωνήσει με βάση την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των συναδέλφων μας και των Αμερικανών ομολόγων μας. Γι' αυτό ακριβώς εξετάζουμε την θεσμική διάσταση και ακριβώς ε, το ζήτημα είναι ποια πτυχή θα μπορούσε να υπάρχει στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ο ρόλος ε, μία τέτοια ε, συνάντηση είναι ακριβώς να έρθουμε σε επαφή και βέβαια να υπάρχει και μια αλληλεπίδραση σε όλα τα υπόλοιπα σημεία της συμφωνίας για να μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να υπάρχει κάτι στην ίδια τη συμφωνία που βοηθάει την αλληλεπίδραση είναι σημαντικό. την είχαμε ήδη συζητήσει, έχει σημειωθεί η πρόοδος για την τρίτη πτυχή που είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό αφορά το τι εργαλεία θα έχουμε για να έχουμε λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς μπορούν να γίνουν εξαγωγές στη ΣΥΠΑ τι απαιτήσει πρέπει να πληρούν τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί ο ρόλος τους στο διεθνές ε, εμπόριο. Λοιπόν, συνεχίζονται οι συζητήσεις, αλλά δεν υπάρχει ακόμα πλήρης συμφωνία για το περιεχόμενο των πληροφοριών και το τι πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για να έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα ε, σε ένα σημείο, ένα site ουσιαστικά όπου θα βρίσκουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Όταν μιλάμε τώρα για την ενέργεια και τις πρώτες ύλες είχαμε δύο ημέρες συζητήσεων στην ενέργεια και τις ε, πρώτες ύλες ε, όπως όπου τονίστηκαν τα ζητήματα που έχουμε συζητήσει στους 10 προηγούμενους γύρους, τα πιθανά στοιχεία που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο κομμάτι του TTIP που αφορά την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Είχαμε λεπτομερείς συζητήσεις και σε ζητήματα τα οποία δεν είχαμε ευκαιρία να συζητήσουμε σε προηγούμενους γύρους π.χ. στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βεβαίως πρόκειται για μια σημαντική πτυχή γιατί θέλουμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για ενέργεια και πρώτες ύλες, αλλά και οι κανόνες που θα συμπεριληφθούν σε άλλα κεφάλαια της συμφωνίας θα ισχύουν για ενεργειακά προϊόντα και επένδυση στον τομέα της ενέργειας. Οπότε η σχέση με το οριζόντιο, με το οριζόντιο κεφάλαιο είναι πάρα πολύ σημαντική πτυχή. Τώρα, με βάση αυτές τις συζητήσεις των δύο ημερών, επαναλάβαμε την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως η TTIP θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες προβλέψεις για την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Εμείς θεωρούμε θα πρέπει να αντιμετωπίζει δύο πράγματα αυτό. Πρώτα απ' όλα τις περιορισμούς εξαγωγών που υπάρχουν στη ΣΥΠΑ για εξαγωγές αργού πετρελαίου και φυσικό αερίου και ένα τέτοιο κεφάλαιο επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και κανόνες ε, που θα ορίζουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ανταγωνιστικό για ζητήματα ενέργειας. Ε, ένα υπόδειγμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικέ διαπραγματεύσεις και θα μπορούσε άρα να συνεισφέρει στον ρόλο της TTIP που είναι η ανάπτυξη παγκοσμίων κανόνων. Η αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να μιλήσει για τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου δεν είναι σε θέση να μιλήσουν για τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου κεφαλαίου λένε πως η απόφαση αυτή θα πρέπει να ληφθεί μετά στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Να σας πω επίσης πως είχαμε όπως ξέρετε και πολλή δραστηριότητα στο Κογκρέσο για ζητήματα ενέργειας που συζητήθηκαν ε, πάρα πολλά νομοσχέδια που είχαν στόχο το να σταματήσει η απαγόρευση εξαγωγής πετρελαίου από τις ΗΠΑ. Ξέρετε πως κάποιοι από αυτούς τους νόμους έχουν προχωρήσει ειδικά στην πλευρά της Βουλής των Αντιπροσώπων ε, έγιναν κάποιες ψηφοφορίες αλλά δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί η γερουσία δεν έχει προχωρήσει ακόμα Ένα άλλο στοιχείο που ήθελα να αναφέρω κύριε Πρόεδρε αφορά τον ε, νομοθετικό διάλογο, τον διατλαντικό νομοθετικό διάλογο που έλαβε χώρα στις 4 Νοεμβρίου στην Ουάσιγκτον και ξέρουμε πως τα ζητήματα ενέργειας και πρώτων υλών είχαν συζητηθεί κατά τη διάρκεια του διατλαντικού ε, ενεργειακού διαλόγου και βεβαίως ε, έγινε και συζήτηση με τον ε, εμπορικό απασταλμένο τον ΙΠΑ και βεβαίως κάποιες άλλες συναντήσεις στο περιθώριο του διαλόγου τέτοιο ζήτημα με χαρά είδαμε πως εκδόθηκε μια κοινή δήλωση που στήριζε ρητός ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την ενέργεια. Αυτό βεβαίως ε, συμφωνεί και με τον διαπραγματευτικό μας στόχο και είναι ενδιαφέρον να δούμε πως ε, με την υιοθέτηση αυτής της κοινή ε, δήλωσης έχουμε και κάποια στήριξη από το Κόγκρέσο. Και βεβαίως είμαστε ευγνώμονες για την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. για τα μηνύματα αυτά που στέλνετε και είμαι σίγουρος πως έχοντας παραστεί στο διάλογο αυτό και στις συναντήσεις που γίνονται στο περιθώριο θα διαπιστώσετε κι εσείς πως είναι δύσκολο να διαπραγματεύεται κανείς με τις Αμερικανικές αρχές. Να σας πω τι θα γίνει στη συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Αναμένουμε την επόμενη συνεδρίαση με την Επίτροπο Μάνστρομ και τον απεσταλμένο για το εμπόριο τον Δεκέμβριο και τον 12ο γύρο του χρόνου. Πιθανότατα τον Φεβρουάριο εδώ στις Βρυξέλλες ακόμα δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία αλλά αυτό αναμένουμε. Και βεβαίως ε, το σκεπτικό εδώ είναι ότι τώρα που από την πλευρά των ΙΠΑ, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, του ειρηνικού ολοκληρώθηκαν, ελπίζουμε να υπάρχει και περισσότερη ενέργεια για να εστιάσουν στην TTIP και να καταλήξουμε στα ζητήματα που είναι στη μέση των διαπραγματεύσεων όπως λέμε για να φτάσουμε στην τελική φάση ελπίζουμε του χρόνου αυτά ήθελα να σας πω σας ευχαριστώ έχω αρκετούς συναδέλφους να ξεκινήσω συνάδελφοι ως συντάκτης και της γνωμοδότησής μας από την Ήτρε στην Ίντα. Θα ξεκινήσω λέγοντας πως επισκέφτηκα την Ουάσιγκτον την προηγούμενη εβδομάδα κάτω από προσκλήσεως ε, του κύριου Άπτεν του Προέδρου της Επιτροπής Ενέργειας και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής ε, Τεχνολογίας συμμετείχα, μίλησα σε πολλές εκδηλώσεις που αφορούσαν τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια στρογγυλή τράπεζα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Επίσης ήμουν συμπρόεδρος με τον Φρέντ Άπτον μια κοινή συνεδρίαση των υποεπιτροπών ενέργειας και αυτό στα πλαίσια του διαλόγου των ε, ε, συνομοθετών. Ε, και στο Κογκρέσο και το κύριο θέμα κατά την άποψή μου και που έθεσα εγώ ήταν το άνοιγμα των αγορών ενέργειας εκτός από τις διαδικασίες TTIP κυρίως για το πετρέλαιο και για το υγροποιημένο αέριο. Είναι πιθανό μετά από την ε, συζήτηση ε, με, την, ε, με τον υπεύθυνο της, με την του, της υπηρεσίας ενέργειας και την κυρία Κατρίνη Νόβελη, η οποία είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπεύθυνη πάλι για θέματα ενέργειας. Είναι γεγονός ότι πριν από, ότι από ένα ε, έφτασε στον 1,5 χρόνο ε, η, η αδειοδότηση, το προθεσμία για την αδειοδότηση, δηλαδή 20, μέρες, 20 μήνες πρέπει να περιμένουν οι εταιρείε πριν ε, πάρουν τέτοια αδειοδότηση. Και αν αλλάξει αυτό, ε, θα ήταν κάτι καλό και επίσης το, η νέα αντιμετώπιση ολόκληρου του, του συνόλου του ζητήματος της αδειοδότησης ε, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το, το Κογκρέσο. Συναντήθηκα με κάποιους ε, ε γερουσιαστές συγκεκριμένα με δύο μέλη τα οποία είναι, ασχολούνται με θέματα εμπορίου και ενέργειας. Ε, συζητήθηκαν λοιπόν πάλι και στα πλαίσια αυτών των συναντήσεων το θέματα της ενέργειας και του LNG και φτάνω στις ερωτήσεις. Πώς θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο για την ενέργεια ε, μπορεί να υλοποιηθεί στην, ε, στις Πολιτείε. Ε, και δεύτερον, η Κομισιόν έχει δίκιο να θεωρεί ότι μπορεί να συμφωνήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε σε σχέση με τα δύο θέματα αυτά για την ενέργεια. Δηλαδή, ερωτώ με ποιο τρόπο ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άνοιγμα των αγορών, ε, άμεσο άνοιγμα της αγοράς υγροποιημένου ε, αερίου. Αυτό συζητήθηκε με τους αρμόδιους φορείς, με τον Υπουργό Εξωτερικών, ίσως μέχρι τα μέσα της επόμενης χρονιάς. Και ένα άλλο ζήτημα, οι, δημόσιες, οι δημόσιοι διαγωνισμοί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ε, είναι πολλές, πολλοί περιορισμοί ε, σε αυτές τις περιπτώσεις που ισχύουν ε, και είναι πολύ ισχυρότεροι σε επίπεδο πολιτιών και όχι σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Πώς θα λυθεί αυτό, πώς θα αντιμετωπιστεί. Ο κύριος Κάριντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, όπως και εκείνη που ρωτήσατε εσείς. Α, όχι, αυτή είναι η δεύτερη. Ας αρχίσω με την πρώτη. Μία πιο γενικόλογη. Τώρα που ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις ε, ε, ε, είπα για την TTIP και τώρα έχουν, ασχολούνται οι πολιτικοί με το κομμάτι του ειρηνικού πλέον. Ε, πώς ε, το βλέπουν, βλέπει η άλλη πλευρά. Δηλαδή, κανονικά τους έχουν λυθεί τα χέρια τώρα και μπορούν να ασχοληθούν αποκλειστικά με αυτή τη συμφωνία. Γιατί ε, η δική μας η συμφωνία δεν έχει θέμα απώλειας θέσεις εργασιών αντίθετα με τον ειρηνικό. Και δεύτερον, εμείς θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο ότι θα ήταν ε, καλό αυτό το κεφάλαιο ε, για τις θέσεις εργασίας. Ε, τι, τι εμποδίζει τους Αμερικανούς, γιατί δεν το δέχονται. Αναρωτιέμαι το ίδιο με εσάς. Ευχαριστώ, συνάδελφος Κόφολ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κεφάλαιο το ενεργειακό. Θέλω να, να σας ρωτήσω κάτι, όχι για τους περιορισμούς για τις εξαγωγές, αλλά για τους κανόνες. Μπορείτε να επεκταθείτε, υπάρχει συνεννόηση με τους Αμερικανούς. Ποιους κανόνες επιδιώκουμε να θεσπίσουμε στο κεφάλαιο για τις ε, πρώτες ύλες, ακατέργας πρώτες ύλες, πρώτη ερώτηση και δεύτερον για τον ενδέκατο γύρο που μας περιγράψατε. Είπατε φυσικά ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η φόρος ανάπτυξη όπως την εννοούμε εμείς είναι ένα θέμα που συζητήθηκε. Ε, οι Αμερικανοί πώς το εκλαμβάνουν όταν μιλάμε για περιβάλλον, εργατικά δικαιώματα, γιατί για μας και αυτά είναι τμήμα του ε, θεμητού ανταγωνισμού. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης για μας Μπορείτε να, μπορείτε να μας ενημερώσετε για αυτό. Για το TLD ε, επειδή ασχοληθήκαμε και το, με το USTR και εγώ ήμουν μέρος της TLD και κάναμε κοινή δήλωση με τους Αμερικανούς για να έχουμε ειδικό κεφάλαιο Γι' αυτό το ρωτάω και στο Κογκρέσο υπάρχει αντίθετη δυναμική δεν, ε, κάποιοι ρεπουμπλικάνοι δεν θέλουν να, δεχτούν αυτή την πράξη, δηλαδή για τις κλιματικές αλλαγές ε, και, ε, δεν υπάρχει συμφωνία με το Κογκρέσο, οπότε υπάρχει περιθώριο κοινή δράσης και μπορεί κάτι τέτοιο ενδεχομένως να συμπεριληφθεί σε μια εμπορική συμφωνία. Ευχαριστούμε, κυρία Νίπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Να σας ρωτήσω τώρα αναφέρατε τα βασικά θέματα το αντικείμενο του 7ου γύρου των διαπραγματεύσεων. Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα ή ενδιάμεσο αποτέλεσμα. Είπατε κάτι για τους δασμούς, αλλά θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο πιο λεπτομερώς. Και έχω και ένα ερώτημα για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Είπατε ποιους κλάδους αφορά. Μπορείτε να μας ενημερώσετε πιο λεπτομερώς. Και τελευταία ερώτηση. Ξέρω πως η προστασία των δεδομένων δεν είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, αλλά το 10 τοποθετήθηκε πρόσφατα για το θέμα αυτό. Μήπως το αναφέρατε έστω στο περιθώριο των συζητήσεων σας. Σας ευχαριστώ. Κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την ε, ενημέρωση. Με ενδιαφέρει το θέμα της ενέργειας ε, και κυρίως το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ε, αναφερθήκατε κι εσείς ε, σε αυτό, Πρόεδρε. Περιμένω την απάντηση που θα δοθεί σε ερωτήσεις σας. Για, το χρονοδιάγραμμα, το Φεβρουάριο έχουμε το 12ο γύρο. Πόσοι άλλοι έχουν προγραμματιστεί και πότε πιθανολογείται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, θα συμπέσουν και με τις αμερικανικές ε, εκλογές επερχόμενες. Πότε εμεί θέλουμε να έχουν ε, ολοκληρωθεί και πόσους γύρους έχουμε ακόμη προγραμματίσει για τα εκκρεμή ζητήματα πέρα από τον 12ο. Και τρίτον, για τις μικρομεσαίες είναι καινούργιο το κεφάλαιο και το καλωσορίζουμε. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες ε, λεπτομέρειες, διότι όσοι είναι θετικά διακείμενοι εδώ στο Κοινοβούλιο αντιμετωπίζουν ε, τα, ε, διαρκώς τα επιχειρήματα όσων είναι κατά και με επιχειρήματα που δεν ευσταθούν. Όμως εμείς δεν έχουμε πληροφορίες για να τα αντικρούσουμε σωστά αυτά τα επιχειρήματα. Και πρέπει να ξέρουμε και τι σημαίνει στην πράξη αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή γενικά για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε θετικές δηλώσεις. Όλο ακούει ο κόσμος ανετικά επιχειρήματα που βασίζονται σε στρεβλές πληροφορίες. Ε, πρέπει να ε, υπάρξει ένα κίνημα με το ε, αντίθετο, δηλαδή με σωστά ευσταθεί επιχειρήματα θετικά. Η κυρία Λόπες Μπερμέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας ε, σε αυτήν τη συνεδρία για να μας πείτε πώς ε, προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Δεν άκουσα καμία αναφορά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτήν την, ε, σε αυτή την συμφωνία κυρίως και μετά από τα όσα συνέβησαν στην Volkswagen. Η υπερβολική συγκέντρωση ε, οδηγεί σε κίνδυνο που διατρέχει η οικονομία να μείνει στα χέρια ε, ορισμένων και λίγων. Το θέμα των εκπομπών ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει δοθεί μεγάλη, μεγάλο σε αυτήν την κατάσταση και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας και τι έχετε να μας πείτε όσον αφορά τον, τα τεστ για τους ελέγχους εκπομπών. Δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε εάν ε, σκοπεύετε να συμπεριλάβετε ε, ρήτρες ε, κοινωνικών ε, στοιχείων για τις δημόσιες προμήθειες και τους δημόσιους διαγωνισμούς και επίσης με ποιο τρόπο θα διευκολύνεται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς που πάντα δυστυχώς μένουν στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων και μια και θέλετε να κάνουμε και κάποιες συστάσεις όσον αφορά τι ε, τις προτάσεις για τον μήνα Φεβρουάριο, ίσως εδώ ε, ε, πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη την εγγύηση της διατήρησης των θέσεων εργασίας, τις ρήτρες, τις κοινωνικές ρήτρες όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τους δημόσιους διαγωνισμούς και τις δημόσιες προμήθειες. Επίσης, όσον αφορά την, ε, την ενέργεια, ε, ε, η, το άνοιγμα, η νέα αντιμετώπιση θα περιλαμβάνει και την υδραυλική ρηγμάτωση και την, το άνοιγμα στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Έχουμε και άλλους ομιλητές στο κατάλογο. Ήθελα μόνο να σας υπενθυμίσω σε σχέση με τα σχόλιά σας ότι στη συζήτηση με τη ΣΥΠΑ για την άρση της ε, διαδικασίας ε, αδειοδότησης. Δεν ζητάμε καμιά χάρη, θέλουμε μια αμοιβαίως υποφελή ε, κατάσταση και τουλάχιστον από τους ρεπουμπλικανούς αλλά και πολλοί δημοκράτες θέλουν να γίνει αυτό και πολλοί γερουσιαστές μας υποστηρίζουν. Δύο ανέφερα ήδη από την Βόρεια Ντακότα και από την Αλάσκα, αλλά και κάποιοι άλλοι ενδιαφέρονται πολύ για την άρση ε, της διαδικασίας αδειοδότησης να ανοίξει η αγορά για τις εξαγωγές. Από, για μας από στρατηγική σκοπιά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, για ο πολιτικός πως επίσης, αλλά και ως προς την τιμή των ενεργειακών προϊόντων. Και στη ΣΥΠΑ και για την Ευρώπη. Αυτά στο... σε σχέση με τα σχόλια σας. Μπορείτε να απαντήσετε και να κάνετε τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για τα διάφορα σχόλια και ερωτήσεις που κάνετε. Θα προσπαθήσω εντάχει να τα καλύψω. Ρωτήσατε αν ε, το κεφάλαιο για τα ενεργειακά προϊόντα και τις πρώτες ύλες είναι δυνατόν. Ναι όχι μόνο είναι δυνατόν κατά τη γνώμη μας, αλλά είναι και ευκταίο και πολύ χρήσιμο θα ήταν να δώσουμε απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις που ε, θέσατε, ενεργειακή ασφάλεια δηλαδή, ανταγωνιστικότητα, των βιομηχανιών με εντατική ε, χρήση ενέργειας, ε, ούτως ώστε τις ενεργοβόρες βιομηχανίες δηλαδή, για να καλύψουμε αυτό το χάσμα που υπάρχει ε, στη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ. Για το κεφάλαιο συγκεκριμένα, έχουμε αφενός το θέμα των περιορισμών των εξαγωγών, σε αυτά που είπατε αναφερθήκατε και σε μέσα που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τους περιορισμούς. Αλλά επίσης θα πρέπει να συμφωνήσουμε για ένα minimum set ε, κανόνων για την ενέργεια και τις πρώτες ύλες. Θεωρούμε ότι χρειάζεται αυτή η δέσμη κανόνων διότι οι κανόνες ΠΟΕ δεν καλύπτουν πλήρως και εξ τον τομέα αυτό και γι' αυτό σε ορισμένες διμερείς συμφωνίες με εταίρους άλλους όπως η Ουκρανία, η Γεωργία, η Μολδαβία έχουμε ήδη αρχίσει ε, την εκπόνηση ειδικών κανόνων για τα ενεργειακά προϊόντα και πρώτες ύλες ε, χρησιμοποιώντας φυσικά και τη δυναμική της TTIP για να ε, εμπλουτίσουμε αυτούς τους κανόνες και να φτιάξουμε ένα τέμπλετ, ένα μορφότυπο που θα μας βοηθούσε να θεσπίσουμε μελλοντικά και παγκόσμιους κανόνες. Μας ρωτήσατε για τις κρατικές προμήθειες ε, και τις δυνατότητες ε, που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ε, σε κυβερνητικό επίπεδο στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ. Όντως, θα πρέπει να εξεταστείτε το ζήτημα όχι μόνο σε ομοσπονδιακό επίπεδο στη ΣΥΠΑ, αλλά και σε επίπεδο πολιτιών. Ξέρετε πως πρόσφατα ε, διαπραγματευθήκαμε με τον Καναδά Προσπαθήσαμε και σε περιφερειακό, κομιτιακό επίπεδο και σε ε, ομοσπονδιακό επίπεδο να το καλύψουμε το ζήτημα και το ίδιο προσπαθούμε και με τη ΣΥΠΑ. Ε, φυσικά η αρχή της εθνικής μεταχείρισης ε, θα πρέπει να εφαρμοστεί γιατί έτσι δημιουργούνται δυνατότητες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν δηλαδή να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για κρατικές προμήθειες και στη ΣΥΠΑ. να, ένας τρόπος με τον οποίο οι μικρομεσαίες θα μπορούσαν ε, να μετάσχουν σε τέτοιες συμβάσεις για ε, κρατικές προμήθειες χάρη σε αυτή την ε, αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τώρα, με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων TPP δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο. Σας είπα ότι ήταν καλός ο γύρο διαπραγματεύσεων με ε, θετικά μηνύματα από πλευρά των ΗΠΑ. Φυσικά, από πλευρά είπα θέλουμε να γίνουν περισσότερες προσπάθειες και τώρα που ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις TPP μπορούν να ασχοληθούν περισσότερο με την TTIP. Ε, βεβαίως χρειάζεται συζήτηση με το Κογκρέσο για την εκείρωση της ε, συμφωνίας, αλλά ούτως ή άλλως ε, οι συμφωνίες, αν δεν είναι, παράλληλες, δεν είναι αντικείμενο παράλληλων διαπραγματεύσεων, φυσικά υπάρχει μεγαλύτερη, περισσότερη ενέργεια και θέληση από πλευρά των Αμερικανών να ασχοληθούν με την TTIP. Κεφάλαιο ERM θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι ένα αντικείμενο διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες ελευθερίου εμπορίου FTA, εκτός από την ναύτα που ε, είναι πολύ παλιά το έχουν αποφύγει σε άλλες διμερείς εμπορικές συμφωνίες ε, για τα, ε, την ενέργεια και τις πρώτες που προσπαθούν να το προσεγγίσουν το θέμα από πλευράς οριζοντίων διατάξεων. Δεν διαφωνούμε, αλλά θεωρούμε πως ε, παρόλα αυτά χρειαζόμαστε ειδικότερε διατάξεις, διότι οι οριζόντιες δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα, ειδικά στον τομέα των ενεργειακών προϊόντων. Και στις συζητήσεις που κάνουμε με τους ομολόγους μας, από τη ΣΥΠΑ, προσπαθούμε να τους πείσουμε για την χρησιμότητα αυτών των ειδικών διατάξεων. Δηλαδή, να έχουμε και κάποιες ε, ε αλλά και κάποιες ειδικέ διατάξεις για τα ενεργειακά προϊόντα, για τα ειδικότερα προβλήματα. Ε, τι άλλο το κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης και αντίδραση είπα, με ρωτήσατε. Περιορισμένη θα έλεγα προς το παρόν. Παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας. Από πλευράς μας είπαμε τι περιέχει συμφωνία. Δεν έχει καταθέσει η αμερικανική πλευρά ακόμη πρόταση, οπότε το θέμα ήταν πιο πολύ διευκρίνηση της πρότασής τους πρόοδος που θα καταθέσουμε. Ε, με ρωτήσατε επίσης ε, τα περί κλιματικών αλλαγών. Φυσικά, εδώ μιλάμε για διαπραγματεύσεις εμπορικού χαρακτήρα. Ταυτόχρονα είναι ξεκάθαρο για μας πως ε, στο μέτρο που συζητάμε και ενεργειακά προϊόντα και πρώτες οι οι διατάξεις θα συμπεριλαμβάνονταν τελικά σε ένα τέτοιο κεφάλαιο ε, που δεν μπορούν να υπονομεύσουν τους στόχους μας ε, για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό το έχουν διευκρινίσει και τα δύο μέρη. Το αντίθετο θα πρέπει να λειτουργούν προς επίρρωση αυτών των στόχων της περιβαλλοντικής μας πολιτικής η τίτλη, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάζει τους στόχου της πολιτικής καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Άλλη ερώτηση σχετιζόταν με την ε, προστασία των ατομικών δεμένων και αν ε, είναι ένα θέμα που καλύπτεται από αυτό το γύρο διαπραγματεύσεων. Όπως ξέρετε δεν είναι ε, τμήμα των συζητήσεων και δεν συζητήθηκε λοιπόν κατά τη διάρκεια αυτού του γύρου. Επίσης, ρωτήσατε Ποιοι είναι οι τομείς όπου έγιναν ειδικότερε συζητήσεις. Ε, υπάρχει μια ομάδα εννέα τομέων που συζητούνται ενδεχομένως για τομεακά παραρτήματα, ε, φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές, ε, ιατροτεχνικές συσκευέ, καλλιντικά, κλωστοϊφαντουργικά, αυτοκίνητα, ε, νέες τεχνολογίες, ε, πληροφορίες, ε, χημικές ουσίες, ζυζανιοκτώνα, μηχανολογία. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι συζητήσει που κάνουμε με τη ΣΥΠΑ για τα αυτοκίνητα σχετίζονται με την ασφάλεια, αλλά σε καμία περίπτωση για τα πρότυπα των εκπομπών δεν συζητάμε, διότι δεν ανήκουν στην ε, στο ρυθμιστικό θεματολόγιο, αν θέλετε, τη είπα. Κατόπιν, ποιος, ε, ποιος είναι ο πιθανός αντίκτυπος της απελευθέρωσης της αγοράς ενεργειακών προϊόντων, με ρωτήσατε, κυρία Λόπες και ε, για την υδρορυγμάτωση πιο θα ήταν ο πιθανός αντίκτυπος επίσης ε, με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, τίποτα μέσα στη συμφωνία δεν μπορεί να επηρεάσει τα κυρίαρχα δικαιώματα κάθε συμβαλόμενου μέρους για τη λήψη απόφασης σε σχέση με το αν πρέπει ή δεν πρέπει να ε, υπάρξει ε, να γίνει έρευνα ή εξόριξη ή εκμετάλλευση οποιοδήποτε ορυκτού πλούτου. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα στην που λέμε μόνο πως εάν τεθεί αυτό το ζήτημα, εν τη αυτή περιπτώσει δεν πρέπει να υπάρξει καμία διάκριση σε σχέση με τη διαθεσιμότητα ε, ε, του ορυκτού πλούτου. Θα τελειώσω απαντώντας και στον κύριο Κέλλη για τις μικρομεσαίες. Δεν έχω αυτή τη στιγμή χρόνο να αναπτύξω περισσότερο το θέμα, αλλά μπορούμε να έρθουμε διμερώς σε επαφή. Για την, το χρονοδιάγραμμα, ο επόμενος γύρος θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο. Συνολικά το 2016 δεν μπορώ να προκρίνω. Να προδικάσω πόσοι θα είναι. Θα προσπαθήσουμε να σημειώσουμε την μέγιστη δυνατή πρόοδο το 2016. Ε, το ιδανικό θα ήταν με την κυβέρνηση Ομπάμα να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Είναι δύσκολο όμως να το προβλέψουμε αυτό. Εμείς σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να προχωρήσουμε με τα mid-game issues, τα επωνομαζόμενα, το 2015 για να ασχοληθούμε με τα end-game issues το 2016. Ε, για να σχηματίζουμε και πιο ξεκάθαρη εικόνα όταν ασχοληθούμε με αυτά τα τελικά ζητήματα ε, σε σχέση με το πέρας των διαπραγματεύσεων. Λέει ο Πρόεδρος, ε, πολύ αργά τώρα για να ξεκινήσουμε νέα συζήτηση. Κύριε Τούρμες, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ζητώ συγγνώμη. Μια πρόταση, μήπως θέλετε να πείτε. Νομίζω ότι το θέμα είναι να δούμε πώς ε, μπορούμε να ανοίξουμε και την ε, αμερικανική αγορά στις ευρωπαϊκές ε, εταιρείες να έχουν περισσότερες ευκαιρίες λοιπόν οι εταιρείες αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Νομίζω πάντως ότι ο ε, καθένας, ο κάθε πολιτικός ε, πρέπει να εξηγεί στους ε, πολίτες του, στους ψηφοφόρους του τι συμβαίνει. Όσο πιο κοντά θα φτάνουμε λοιπόν στις εκλογές, τόσο πιο δύσκολες θα γίνονται οι συζητήσεις από την Αμερικανική πλευρά που έχει μπροστά τις εκλογές. Άρα πόσο χρόνο έχουμε μπροστά μας πριν ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα καθαρά πολιτικό ερώτημα. Ζήτησα, ε, έκανα την ίδια ερώτηση σε όλους τους Αμερικανούς. Πώς θα πείσετε την ε, ε, δημόσια την κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς θα πείσουμε την κοινή γνώμη στην Ευρώπη για το TTIP και την αξία του. Είναι πολιτική ερώτηση και έχετε δίκιο από την υποβάλλατε. Λοιπόν, να σας πω ότι ε, οι συντονιστές πήραν τις ε, εξής αποφάσεις. Ε, συνεκτική πολιτική για την καινοτομία θα το αναλαμβάνει το ΕΛΚ. 2 μελέτη για την ε, έρευνα, για την αντίκτυπο στην αγορά όσον αφορά τη ρομποτική και την ψηφιοποίηση. Πέτρα ε, είναι εκπρόσωπος της ε, Ήτρε και ο Σλάνσκος Αντάλγας ορίστηκε αναπληρωτής. Σημείο 3 οι συντονιστές αποφάσισαν να ξεκινήσουν την ε, paperless ε, πρωτοβουλία από τον Ιανουάριο του 2016. Ε, επομένως, μάλλον ατομικά θα ειδοποιηθούν τα μέλη της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Σε δύο μήνες από τώρα θα αρχίσει να ισχύει το paperless. Επίσης, αποφάσισαν ε, οι εισηγητές ότι οι συμβαστικές τροπολογίες θα είναι πλέον διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά. Βεβαίως μπορεί κανείς να διαμαρτυρηθεί αν θέλει, αλλά εάν διαμαρτυρόμαστε δεν θα είμαστε ποτέ έτοιμοι στην ώρα μας. Ε, η πολυγλωσία είναι καλό πράγμα και πολύ σημαντική για όλους μας, αλλά η απόφασή μας, η απόφαση των συντονιστών λέει ότι μόνο στα αγγλικά. Τρεις η ώρα κοινή συνεδρίαση ΙΜΚΟ Ήτρε. Τρεις, οκλοκ, ε, ακριβώς παρακαλώ. Είναι σημαντικό να είστε στην ώρα σας. Ε, γιατί έχουμε... Α, να σας πω... 30 ε, Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου, 30 Νοεμβρίου απόγευμα και 1η Δεκεμβρίου πρωί και απόγευμα η επόμενη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες. Στις 3 λοιπόν κοινή συνεδρίαση ΙΜΚΟ Ήτρε θα τα πούμε λοιπόν σε 2,5 ώρες.